κατάλογο των ε, τρίτων χωρών που έχουν απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης πρώτα απ' όλα η Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Μπαρό, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και λυπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την άρση της βίζας για τα Δυτικά Βαλκάνια. Γι' αυτό οδηγηθήκαμε στη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ όλους όσους με βοήθησαν και το Συμβούλιο και την Κομισιόν για την καλή συνεργασία που είχαμε και αποτελεί καλή βάση για την περαιτέρω συνεργασία στον τομέα αυτών, ειδικά μετά την θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Η δε υποχρέωση για θεώρηση των διαβατηρίων είχε απομονώσει τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων επί σειρά ετών. Οι νέοι άνθρωποι από τις χώρες ε, των Δυτικών Βαλκανίων γνωρίζουν λίγα πράγματα για την Ευρώπη όσα και για την Αμερική. Ξέρουν την Ευρώπη μόνο από το ίντερνετ και την τηλεόραση. Επειδή δεν προέρχομαι από την Σλοβενία πρέπει να πω πως ε, η Σλοβενική Προεδρία το 2008 ξεκίνησε τη διαδικασία απελευθέρωσης της ε, Βίζας. Χαιρετίζω λοιπόν την πρόταση της Κομισιόν για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για Σερβία, Μαυροβούνιο και την Πουγουδομού έτσι ώστε οι πολίτες αυτών των κρατών να μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα και μάλιστα από τις 19 Δεκεμβρίου. 1η πρώτου 2010 έχουμε ένα μεγάλο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί γιατί ακριβώς πολλοί πολίτες αυτών των κρατών θέλουν να ταξιδέψουν για τις γιορτές στην Ευρώπη και η απελευθέρωση βεβαίως ε, θα ενισχύσει και την περιφερειακή συνεργασία και τις ε, πολιτιστικές ε, και κοινωνικές ανταλλαγές. Αγαπητοί συνάδελφοι, η απελευθέρωση τριών χωρών από την υποχρέωση βίζας είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Πρέπει όμως να βοηθήσουμε και άλλες χώρες ε, που δεν έχουν ακόμα απαλλαγή από την βίζα. Πρέπει να δώσουμε και στι χώρε αυτές την δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό το καθεστώς μόλι βεβαίω πληρώσουν αυτά τα κριτήρια. Μιλάω για την Αλβανία και τη Βοσνία Ριζεγοβίνη η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη καθώς θα μπορούν να ταξιδεύουν γρήγορα χωρίς προβλήματα στις γειτονικέ χώρες. Πρέπει να στείλουμε λοιπόν ένα σαφές μήνυμα στις χώρες αυτές. Πρέπει να εργαστούν οι κυβερνήσεις τους και να πούμε πως δεν ε, χρειάζεται και εμείς να επιβάλλουμε ε, περί εμπόδια. Η πρόταση αυτή έχει την στήριξη και της Επιτροπής ε, Εξωτερικών και της δικής μου Επιτροπής, Επιτροπής Ελευθεριών. Αύριο θα ζητήσω τον λόγο ξανά και θα υποβάλω μια πρόταση για απαλλαγή από βίζα των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Θα ψηφίσουμε αύριο την πρότασή μου αυτή και ειδικά για την απαλλαγή της Σερβίας ε, του Μαυροβουνίου και της ε, Πουγουδουμού από 19 Δεκεμβρίου και θα ψηφίσουμε επίσης ε, για την απαλλαγή από βίζα της Αλβανίας και της Βοσνίας Ριζεγοβίνης στο συντομότερο δυνατόν. Θα ήθελα να έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία και για την Αλβανία και Βοσνία Ριζεγοβίνη, αλλά γνωρίζω πως ε, δεν είναι απλές οι διαδικασίες και γνωρίζω πως ε, θα πρέπει να τεθεί ενισχύ η απελευθέρωση μέχρι το καλοκαίρι. Και δεν μην ξεχνάμε και το κοσμοπέδιο. Mm. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την πολιτική ευθύνη να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία και αναμένω ευρεία στήριξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ κύριε Κορατσαβή, έχετε ε, θέμα της διαδικασίας. Ναι, η Σουηδική Προεδρία φαίνεται ότι δεν εκπροσωπείται εδώ σε επίπεδο Υπουργού όπως θα θέλαμε. Από ό,τι έμαθα δεν έχουν προσκληθεί. Τους είπαν ότι δεν χρειάζεται η παρουσία της. Θα υπενθυμίζω όμως ότι η Σουηδική Προεδρία έχει θέσει πρώτη το θέμα της κατάργησης των θεωρήσεων. Και η συνάδελφός μου Τάνια η συγγήτρια θα συμφωνεί. Θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε γιατί τους χρωστούμε την κοινή δήλωση που έγινε από Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και με υποστήριξη της Κομισιόν που είναι μοναδική στην ιστορία του οργάνου εδώ. Θα ήθελα λοιπόν να μου δοθεί μια εξήγηση, όχι τώρα και εδώ, αλλά να γραφτεί στα πρακτικά ότι δεν προσήλθε ο Υπουργό γιατί δεν προσεκλήθη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με ευχαριστώ. Με πληροφορούν πως η Προεδρία του Συμβουλίου προσεκλήθη αλλά υπήρχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις. Γι' αυτό απουσιάζει. Παρακαλώ, κατόπιν τον λόγο τώρα έχει η Κομισιόν, ο κύριος Μπαρό. Ευχαριστώ. Όντως, όπως είπε η κυρία Μπίλτ, η Ισουδική Προεδρία ήταν εξαιρετικά δραστήρια στον τομέα αυτό. Γιατί θέλει, όπως και εμείς, να δώσουμε νέες δυνατότητες στους πολίτες και ιδιαίτερα στους νέους για κινητικότητα, να γνωρίσουν καλύτερα την Ευρώπη μας. Είναι λοιπόν μια ιστορική καμπή στην ανάπτυξη της Ευρώπης η κατάργηση των βραχυπρόθεσμων θεωρήσεων. Όλοι γνωρίζουμε την ευαισθησία του ζητήματος που αφορά όλους τους πολίτες των συγκεκριμένων χωρών. Κατανοώ βεβαίως τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα στα πλαίσια αυτά να επανεβιβαιώσω την βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρακολουθήσει εκ του σύνυγκης την εφαρμογή όλων των κριτηρίων που έχουν συμπεριληφθεί στον λεγόμενο οδικό χάρτη ή αλλιώς φύλλο Για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είχαμε κάνει μια εμπειρογνωμοσύνη τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα για τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Κάναμε αποστολή τον Οκτώβριο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, αποστολές που επιβεβαίωσαν ότι όλα τα κριτήρια του φύλου πορείας των αντιστοίχων φύλων πορείας για κάθε χώρα δηλαδή έχουν εφαρμοστεί σωστά. Για την Αλβανία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη θα ακολουθήσουμε την ίδια μέθοδο. Παρά σημαντικές προόδους που έλαβαν χώρα τους τελευταίους μήνες, η Βοσνία και η Αλβανία δεν μπόρεσαν ακόμα να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που πρεσβεύει το φύλλον πορείας και που να δικαιολογούν την κατάργηση της υποχρεώσεως βραχύπροθεσμης θεώρησης. Όπως είπε μια συνάδελφος, ευρωβουλευτής, αποτελεί για τις χώρες αυτές μεγάλη ενθάρρυνση το γεγονός ότι οι γείτονές τους επέτυχαν την κατάργηση της βραχυπρόθεσμης θεωρήσεως και είμαι σίγουρος ότι θα θελήσουν και η Αλβανία και η Βοσνία να κάνουν παν δυνατό για να επιτύχουν το αυτό. Καλό το Κοινοβούλιο να συνομοθετήσει στον τομέα αυτό, διότι με την θέση σε ισχύ της ε, συνθήκης της Λισαβόνος είναι απαραίτητη η συνομοθετική δραστηριότητα του Κοινοβουλίου. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα δημιουργούσε σύγχυση και δεν θα επέφερε μια πραγματική αλλαγή στο καθεστώς των θεωρήσεων. Θα δημιουργούσε πλαστές, κύβδηλες, φρούδες ελπίδες σε σχέση με αυτά που απαιτεί το φύλλον πορείας. Η Αλβανία και η Βοσνία μπαίνουν στο παράδειγμα ένα του κανονισμού προς το παρόν και επανεπιβεβαιώνουμε ότι αυτή τη πληρώσουν τα κριτήρια δύο χώρες αυτές θα μπορέσουν να απολάβουν του μέτρου της κατάργησης, της θεώρησης και αυτές. Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει το κείμενο της πολιτικής κοινή δήλωση όπου επιβεβαιώνει την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσει σε ισχύ το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, κατάργηση των θεωρήσεων για τους πολίτες της Αλβανίας και της Βοσνίας Ερκοβίνης όσο το δυνατόν πιο σύντομα υπό την προϋπόθεση όπως είπα προηγουμένως ότι οι χώρες αυτές ε, θα προβούν στα βήματα που ακόμα δεν έχουν κάνει. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η Βαρόνι Λάντφορτ για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η δέσμευση που υποστηρίζεται στην τελική έκθεση και από την δήλωση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου είναι μια δέσμευση που βλέπει στο μέλλον. Δεν είναι καθαρά αλτρουιστική η κίνηση αυτή απελευθέρωσης από την Βίζα, καθώς είναι μια έξυπνη κίνηση. Θα προωθηθεί η ασφάλεια με την ευρύτερη έννοια. Οι ελεύθεροι άνθρωποι, οι άνθρωποι που ταξιδεύουν συνήθως αναζητούν ειρηνικές λύσεις και δεν είναι εσωστρεφείς και εθνικιστές, κάτι το οποίο αποτελεί κίνδυνο ασφάλειας. Ποιος δεν συγκινήθηκε από τις εικόνες και τους πανηγυρισμούς που είχαμε αυτή την εβδομάδα για την 20η ε, επέτειο από την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Βεβαίως αυτά τα εμπόδια δεν συγκρίνονται με το τείχος του Βερολίνου, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδια για την ελεύθερη εκείνη των ανθρώπων, την αμοιβαία κατανόηση και την ανεκτικότητα. Οπότε θα πρέπει να διασφαλίσουμε δίκαια αποτελέσματα 15 χρόνια μετά τη συμφωνία του Ντέιτον. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για τη σκληρή της δουλειά και για το πώς συμπεριέλαβε όλους και οδησυγητές δύσκολη αυτή η πορεία τους τελευταίους μήνες. Να ευχαριστήσω το Συμβουλίο και ειδικά τη Σουηδική Προεδρία για το έργο της, για το πώς μας βοήθησε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για την δήλωση που καθορίζει τον οριστικό στόχο απαλλαγής από βίζα για όλους τους πολίτες των Δυτικών Βαλκανίων του νομότερο δυνατόν και ελπίζουμε αυτό να γίνει το 2010 γιατί ε, η κατάσταση διαιρεί και δημιουργεί αστάθεια το να μην υπάρχει δηλαδή μια κίνη λίγο πολύ ημερομηνία για να μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα και δεσμευτήκαμε επίσης στην έκθεση φαγιών να εργαστούμε για διευκόλυνση και απελευθέρωση ε, του καθεστώτος για το κοσφοπέδιο ε, σε χρονοδιάγραμμα παρόμοιο με τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Επίσης, να προσθέσω την ελπίδα μου, να εκφράσω την ελπίδα μου, ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν είναι στην ζώνη Σέγγεν ακόμα θα ακολουθήσει σύντομα στον ίδιο δρόμο. Υπάρχει μια σχιζοφρένεια για μένα να εργάζομαι στα ζητήματα Σέγγεν γιατί είμαι Βρετανίδα Ευρωβουλευτής. Αλλά προφανώς καλό θα είναι και για την Ευρωπαϊκή Ανδυτικά Βαλκάνια να ακολουθήσει και το Ηνωμένο Βασίλειο των Συντομότερων να τελειώσω ευχαριστώντα ξανά την κυρία Φαγιών την εισηγητρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στου ομιλητέ εξ ονόματο των ομάδων. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ για δύο λεπτά για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Είμαστε αποφασισμένοι να επιταχύνουμε τη διαδικασία κατάργησης των βυζών μέχρι τον Ιούλιο του 2010. και να καταργηθούν οι θεωρήσεις για τη Σερβία, τη Βοσνία και το Μαυροβούνιο μέχρι τα Χριστούγεννα. Κατανοούμε βέβαια την έκκληση των λαών της Αλβανίας και της Βοσνίας. Είναι μια νέα γενιά η οποία έχει κλειστεί στη χώρα της και δεν μπορεί να βγει χωρίς θεώρηση. Πρέπει να τους δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να τους δεχτούμε. Είναι λυπηρό ότι μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει τέτοια εξέλιξη γιατί τις καθυστερήσεις τις έκαναν οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών και όχι εμείς. Εμείς τους ζητήσαμε να εφαρμόσουν τα κριτήρια όσο το δυνατόν συντομότερα και ξέρουμε ότι η Κομισιόν βοηθάει σε αυτό. Κυρία Πρόεδρε, δυστυχώ αναγκάζομαι να εκφράσω τη λύπη μου γιατί χρειάστηκαν τρεις μήνες διαπραγματεύσεων για να πιστεί η αριστερά του Κοινοβουλίου από το ΕΛΚ τι να κάνει να εφαρμόσει τις συνθήκες. Δεν είναι το δύσκολο πράγμα. Δεν ήταν. Τέλος το κατάλαβαν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι υπεράνω του νόμου και με όλο το σεβασμό που οφείλω στους διακεκριμένους συναδέλφους μου πρέπει να τους δηλώσω ότι η στάση τους δεν ήταν επικοδομητική. Δεν υπάρχουν εδώ μαγικά. Τελεία. Ούτε είμαστε εδώ σε αγώνα. Είναι, είμαστε εδώ για να έχουμε απτά αποτελέσματα για τους πολίτες των Μπαλκανίων. Θα ήθελα να είμαι σαφής. Οποιοδήποτε, οποιοδήποτε προσωρινό και ανάμεικτο καθεστώς δεν βοηθάει κανέναν και δεν, στέλνει, δεν αποτελεί καμία πολιτική χειρονομία. Θα ήθελα να καταλήξω λέγοντας ότι αφήστε με να σας το πω παρακαλώ ότι η πολιορκία του Σεράγεβου και ο βομβαρδισμός του είναι κάτι που με έπεισε να τις κόβουν το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μωράης κατόπιν για 1,5 λεπτό από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς. Τους ε, Σοσιαλδημοκράτες, με συγχωρείτε το 2008, από το 2008 και μετά, μετά τη Σλοβενική Προεδρία δεν έγινε μεγάλη πρόοδος για κάτι που σωστά χαρακτήρισε ως ιστορική καμπή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλώ για την κατάργηση των θεωρήσεων. Εκ μέρους των σοσιαλιστών και δημοκρατών θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φαγιό για την κουραστική και αποτελεσματική εργασία της που συνεισφέρει στην κατάργηση του καθεστώτος θεωρήσεων για όλες τις χώρες των Δυτικών ε, Βαλκανίων. Με τους Σκιώδης, με την Κομισιόν, με το Συμβούλιο έγινε αυτή η δουλειά και όλοι αξίζουν εύσημα. Είναι εποφελές μέτρο για όλες τις πλευρές και βεβαίως είναι θέμα και σωστής εφαρμογής του φύλου πορείας σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτές οι χώρες ούτως ώστε το καθεστώς κατάργησης των θεωρήσεων να καταστεί μια επιτυχία. Είναι σωστή η διαπραγμάτευση της Κομισιόν. Η δήλωση που προέκυψε ισχύει για την Μακεδονία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Η Αλβανία και η Βοσνία Ερζεγοβίνη μπαίνουν προ το παρόν στο παράρτημα και ελπίζουμε ότι γρήγορα και αυτές θα συμπεριληφθούν στις άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Λούνατσα και ένα λεπτό για τους πρασίνους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες, να συγχαρώ τις δύο εισηγήτριες ε, για τις Επιτροπές Εξωτερικών και ελευθεριών. Πραγματικά νομίζω πως κατάφερα να κάνουν μια πρόταση και ζητούν από Κομισιόν και Συμβούλιο να κάνουν συνολικό πακέτο για όλους τους ανθρώπους των Δυτικών Βαλκανίων και να μην αφήσουν κάποιους απ' έξω και ελπίζω και απευθύνομαι εδώ στον κύριο Μπαρό ελπίζω εσείς να καταφέρετε να επιβάλλετε στο Συμβούλιο να υπάρξει στόχος απελευθέρωσης και για το κοσφοπέδιο και για τη Βοσνία και την Αλβανία το αργότερο του χρόνου να επιτευχθεί η απελευθέρωση. Εγώ θα ήθελα και νωρίτερα να ξεκαθαρίσω κάτι. Βεβαίως μιλάμε για την εφαρμογή, αλλά ακούσαμε στη Σερβία π.χ. ότι δεν εφαρμόζονται τα πάντα. Πώς το εκτιμάτε. Πρέπει να εφαρμόζονται τα πάντα. Νομίζω είναι σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ τελειώστε, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ λοιπόν όλους όσους συνεργάστηκαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πακ. Δύο λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από 20 χρόνια οι συμπατριώτες μου από την Ανατολική Γερμανία απέκτησαν το δικαίωμα να ταξιδεύουν ελεύθερα και λίγα χρόνια μετά ο Μιλόσεβιτς αυθαίρετα κατάφερε να καταργήσει το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης των ανθρώπων και της Σερβίας και των γειτονικών χωρών και ακούμε εδώ πέρα τις συζητήσεις να, ε, για το πόσο σημαντική είναι η απαλλαγή από βίζα των ανθρώπων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και ξέρουμε πως δεν γίνεται τίποτα εάν δεν συμφωνήσουν οι κυβερνήσεις. Δεν πρέπει να φοβούνται οι λαοί μα. Οι εγκληματίε δεν χρειάζονται καμία βίζα, περνάνε ούτω ή άλλω τα σύνορα. Μιλάμε για τη νέα γενιά η οποία θα επωφεληθεί από την απελευθέρωση τη βίζα και μπορεί επιτέλου να ταξιδέψει όπου θέλει. Χαιρόμαστε λοιπόν για το ότι οι πολίτες ε, Σερβίας, Μαυροβουνίου και Μακεδονίας μπορούν να ταξιδέψουν. Οποία χαρά! Και βεβαίω με θλίψη ακούμε πω ε, Αλβανία, Βοσνία και Κοσμοπέδιο δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμα. Αναμένουμε όμω από την Κομισιόν να μα πει το Δεκέμβριο να διαπιστώσει και να τιμήσει τη μεγάλη πρόοδο τη Αλβανία και να πει πω έχει βελτιωθεί λίγο η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Δυστυχώ στη Βοσνία Ερζεγοβίνη υπάρχουν πολιτικοί που δεν ενδιαφέρονται για του πολίτε του και έχουν μόνο εκείνη απαλλαγή από βίζα. Ελπίζω λοιπόν να επιτευχθεί αυτό για αυτές τις χώρες το επόμενο καλοκαίρι. Δεν ξεχνάμε όμως και το κοσφοπέδιο. Δεν επιτρέπεται να παραμείνει μαύρη τρύπα στο χάρτη. Έχουμε την υποχρέωση να βοηθήσουμε το κοσφοπέδιο να εκπληρώσει τους όρους. Από μόνο του δεν μπορεί. Κυρίες και κύριοι, πρόκειται για ένα ζήτημα καθαρά ανθρώπινο και χαιρόμαστε για το ότι είμαστε σε θέση να το προσφέρουμε σε ανθρώπους. Ευχαριστώ κύριε Μαρό. Ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Γκέντς, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε ως ένα έργο οικοδόμησης της ειρήνης και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως ε, η ενσωμάτωση μπορεί να αποτελέσει πολύ αποτελεσματικό μέσο της ειρήνης και τώρα έχουμε εμεί αυτό το μέσο στα χέρια μας όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια. Τα Δυτικά Βαλκάνια πέρασαν έναν μεγάλο πόλεμο και Τώρα πρέπει να κάνουν βήματα προς τα εμπρός και ένα σημαντικό μέσο για να τους βοηθήσουμε είναι η απαλλαγή από την ε, βίζα και οι προλαλήσαντες ανέφεραν πόσο σημαντικό είναι αυτό για τους νέους ανθρώπους να έχουν τη δυνατότητα δηλαδή να ταξιδέψουν και είναι ένα μήνυμα εμπιστοσύνης το να απαλλάξουμε αυτές τις χώρες από την Βίζα και ταυτόχρονα αυτές οι χώρες θα προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σημαντικό και από πλευράς πολιτικής ασφάλειας και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ε, πρέπει να ξεπεράσουμε τον διχασμό σε αυτή την περιοχή. Ο κύριος Μπουσουτήλ δεν είναι εδώ, τα ακολουθεί η κυρία Μποζκούρτ για ένα λεπτό. Αύριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει για την κατάργηση βίζας για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, όχι όμως για όλες τις ε, χώρες από 1η Ιανουαρίου. Είναι πάρα πολύ ατυχές το ότι ως αποτέλεσμα της τοποθέτησης της Ευρωπαϊκής ε, ε, Επιτροπής θα υπάρχει πρόβλημα με την Βοσνία Ζεγοβίνη μπορούν και θα έχουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί οι οποίοι έχουν διαβατήριο της ε, Κροατίας ή της Ευβίας και μπορούν να ταξιδέψουν και οι λοιποί, δηλαδή οι Βόσνοι μουσουλμάνοι. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτό το δικαίωμα και για τη Βοσνία και για την Αλβανία βέβαια στα κριτήρια είναι κριτήρια όταν μιλάμε για απελευθέρωση από την ε, Βίζα και πρέπει να εκπληρωθούν αλλά θεωρούμε πως όταν εκπληρωθούν πρέπει να υλοποιηθεί η απελευθέρωση το συντομότερο δυνατόν, ειδικά όταν καταβάλλεται τόση προσπάθεια για να εκπληρωθούν αυτά και ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπαρασταθεί σε αυτές τις χώρες για να τα καταφέρουν σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζόραν Τάλερ για 1,5 λεπτό. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η κατάργηση των θεωρήσεων για τους πολίτες των Δυτικών Βαλκανίων είναι τεχνικό μεν θέμα αλλά και πολιτικό. Το συζητούμε μάλιστα σήμερα που γιορτάζουμε την πτώση του τείχους του Βερολίνου πριν από 20 χρόνια. Στην Ποντγκόριτσα, στο Βελιγράδι, θα έχουν ένα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο δώρο. Θα ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση. Ενώ εδώ και πολλά χρόνια ένας τείχος χώριζε τα Δυτικά Βαλκάνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούσαν να διακινηθούν ελεύθερα προς την Ένωση οι πολίτες τους, όπως στην πρωινή Κοσλαβία. Αυτή η απομόνωση είχε ικτρά αποτελέσματα και καιρός ήταν να λήξει πια η περίοδος αυτή. Η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Φυρώμα θα επωφεληθούν από την κατάργηση αυτή και ελπίζω σύντομα και η Βοσνία και η Αλβανία. Πρέπει να μπορούν οι πολίτες των χωρών αυτών να γνωρίσουν την Ευρώπη καλύτερα, να ταξιδεύσουν και να προετοιμαστούν καλύτερα και για τη μελλοντική τους ένταξη. Εγώ είμαι εισηγητής για την Πουγουδουμού και λαμβάνω πολλές τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα και με ρωτάνε όλοι πότε θα ταξιδεύουμε ελεύθερα. Είναι πολύ μεγάλο βήμα προς την Ένωση. Και έτσι η πρώτη ομιλήτρια κυρία Γκάλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και τους κοιόδης εισηγητές να πω το εξής. Σήμερα την επέτειο της πτώσης του τείχους του Βερολίνου είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ε, χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να πέσει και αυτό το τείχος. Γι' αυτό χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία αυτή αλλά το θέμα δεν είναι μόνο τεχνικό. Πρέπει να στείλουμε και ένα πολιτικό μήνυμα. Υποστηρίζω την κοινή ε, δήλωση γιατί έτσι εκφράζουν τα θεσμικά όργανα πως έχουν συνέστηση των υποχρεώσεών τους ε, και θα ανταποκριθούν σε αυτές. Οι ενδιαφερόμενες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει από την άλλη να εκπληρώσουν και αυτές τις υποχρεώσεις τους. Σας ευχαριστώ κύριο Φως. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω πως με τις χώρες των Βαλκανίων είμαστε σε καλό δρόμο, έχουμε προσέγγιση μέσω της διευκόλυνσης της βίζας, οδηγούμαστε σε μια σταθερότητα, δημιουργείται επίσης και μια, κάποιοι, δημιουργείται κάποιες κοινέ αξίες. Πρέπει όμως να έχουμε σαφείς κανόνες και να πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις ε, και να τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις. Βεβαίως ανέφερε και η κυρία Κορατσαμπίλτ πως έκανε αρκετές προσπάθειες. Διαφορετικά νομίζω πως ε, θα απομακρυνθούμε από το σύστημα που έχουμε που είναι σαφές και δεν είναι τίμιο αυτό ούτε για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ούτε για τους δικούς μας τους λαούς τα πολιτικά μηνύματα δεν ε, κολλάνε σε έναν αστερίσκο ή ε, σε μια ευρωπαϊκή οδηγία. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Λουκατσεύσκα έχει κατόπιν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που οι πολίτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων θα μπορούν να διακινούνται ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αυτό θα διευκολύνει τις επαφές μεταξύ ανθρώπων και λαών αλλά και εμπορευομένων. Δεν πρέπει οι ανατολικοί γείτονέ μας να παραμείνουν απομονωμένοι και δεν πρέπει να τους στερήσουμε τις δυνατότητες που δίνουμε σε άλλους. Πρέπει βέβαια να θέσουμε και σαφή κριτήρια στο φύλλο πορείας τους για την ένταξη, διότι για τους ε, λαούς της Ανατολικής Ευρώπης θα χρειαστεί πολύ καιρό μέχρι την ένταξη και εντωμεταξύ πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Το 2012 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα διοργανωθεί από κοινού από την Πολωνία και Ουκρανία και αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντική η της διακίνησης. Ευχαριστώ κύριο Πρέντερ κατόπιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ να τονίσω πόσο ελεύθερη είναι η ελευθερία κίνηση των ανθρώπων είναι θεμελιώδες δικαίωμα και να τονίσω πως πάρα πολλοί πολίτες από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα χαρούν για αυτό το δικαίωμα, γι' αυτό χαιρετίζω αυτή την εξέλιξη. Ταυτόχρονα όμως θέλω να υπενθυμίσω πω η έκθεση αυτή δεν λέει τίποτα για τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης και συγκεκριμένα για την Μολδαβία. Εκεί πέρα έχουν γίνει ε, σημαντικά βήματα στην πολιτική και πρέπει να αναφερθούν. Νομίζω ότι το ψηλότερο τείχος στην Ευρώπη είναι μεταξύ Ρουμανίας και Μολδαβίας και είναι κάτι λυπηρό. Σας ευχαριστώ. Αυτοί ήταν οι ομιλητές στη διαδικασία και Τώρα έχει τον λόγο πάλι η Κομισιόν. Κύριε Μπαρό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές που υποστήριξαν θερμά, τολμώ να πω, την διαδικασία καταρρήσης των θεωρήσεων για τις τρεις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Είπατε όλοι ότι η ελευθερία κίνησης και κυκλοφορίας είναι απόλυτα ευκταίη όπως είπε ο κύριος Μωράης, είναι αποφελής και για τα δύο μέρη, και για αυτές τις χώρες και για την Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώντας όλους τους ομιλητές και την εισηγήτρια πρόφανος, θα ήθελα λέγω να αναφέρω ότι δεν εφίσθημεν προσπαθειών από τότε που ελήφθη η προσπάθεια η απόφαση συγγνώμη, να βοηθούμε ε, την Αλβανία, τη Βοσνία Ερζεγοφίνη για να προοδεύσουν. Και θα συνεχίσουμε να πράττουμε το αυτό. Θεωρώ ότι η ταχεία έγκριση αυτού του ψηφίσματος αποτελεί θετικό ιονό για την μετάγγιση αυτής της διαδικασίας και στις άλλες χώρες, Βοσνία, Ζεγοβίνη και Αλβανία, χωρίς βεβαίως να ξεχνούμε και το Κόσοβο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η εισηγήτρια για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε ακόμη μια φορά για όλα όσα κάνατε και που αποδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την κατάργηση των θεωρήσεων για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Λυπούμε γιατί δεν είναι εδώ η Σουηδική Προεδρία, γιατί η συνεργασία μας ήταν άψογη. Δέχομαι επίσης τη δέσμευση της Επιτροπής που θα κάνει ό,τι μπορεί για να επιταχυνθεί η διαδικασία και για τη Βοσνία και την Αλβανία. Και θα ήθελα και οι δύο αυτές χώρες να υποφελθούν από το καθεστώς απελευθέρωσης των θεω... κατάργησης των θεωρήσεων ίσως και το επόμενο καλοκαίρι. Γνωρίζω πολύ καλά τι προβλέπουν οι συνθήκες, αλλά εδώ είμαστε σε πολιτικό όργανο και θέλουμε να ασκήσουμε την πολιτική σοβαρά. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι χαίρομαι για την κατάργηση των θεωρήσεων για τη Μακεδονία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο από το Δεκέμβριο ήδη και θα ήθελα και η Βοσνία και η Αλβανία να ακολουθήσουν όσο το δυνατόν σύντομότερα γιατί εδώ μιλάμε για την τύχη της νέας γενιάς και είναι πολιτική μας ευθύνη να το λήξουμε αυτό το θέμα, να καταργηθούν οι θεωρήσεις και να βρούμε μια λύση και για όλους τους πολίτες του Κωσυφοπεδίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Φαγιό. και τώρα για αυτό το θέμα εδώ. Θα ψηφιστεί αύριο στις 11 περίπου. Επόμενο θέμα. Επόμενο θέμα. Είναι προφορική ερώτηση για